Οπότε το διευρυμένο Προεδρείο θα γίνει σήμερα το πρωί από τις 11 και μετά. 11 και μισή και μετά. Ο κύριος Παντζέρη σήμερα το απόγευμα και η κυρία Γκόμες που είναι η συγγήτρια για τη συμφωνία με τη Λιβύη και ο κύριος Παντζέρη που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας του Μαγκρέμ, θα έρθουν να μας παρουσιάσουν τα σχετικά. Θα παραταθεί η συνεδρίαση δε σήμερα μέχρι τις 7.30 γιατί θα έρθει ο Επίτροπος ο κύριος Φίλε ο οποίος θα έρθει να μας μιλήσει για την διεύρυνση και για τις υποψήφιες χώρες ή για τις ενδυνάμει υποψήφιες χώρες. Αυτή η συνάντηση θα γίνει μετά το πέρας της συνεδρίαση του Κολεγίου του, του, Σώματος των Επιτρόπων που θα συζητηθεί αυτό το πακέτο. Λοιπόν, έγκριση των πρακτικών της 20 Σεπτεμβρίου 2010 και 5 Οκτωβρίου 2010. Καμία ανακοίνωση του Προέδρου. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Οι συνάδελφοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε ένα ρεκόρ τροπολογιών, 423 τροπολογίες. Και εν ώψη της απογευματινής ψηφοφορίας, Έχουμε καταλήξει σε πολλές συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες. Αυτό θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε στην κυρία Άστον τις ε, θέσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο φυσικά βέβαια να περάσει η έκθεση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου με μεγάλη πλειοψηφία. Η κυρία Αντρική ναι, έχει παρουσιάσει 40 συμβιβαστικέ τροπολογίες. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια να μας παρουσιάσει και τις τροπολογίες αλλά και τις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες καταλήξαμε. Διαδικαστικό? Α, όχι. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Η εισηγήτρια λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα την έκθεση αυτή για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Το κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι το, η κύρια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο δυο παρατηρησει παρατηρήσεις. 2008-2009. Υπήρχε σημαντική ε, εξέλιξη. Θα ήθελα να σας ε, τονίσω καταρχήν ότι καλύπτεται μεγαλύτερη χρονική περίοδο από ό,τι συνήθως από τα μέση 2008 έως τα τέλη του 2009 και καλύπτει όχι μόνο την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ανά τον κόσμο, αλλά και την πολιτική της Ένωσης και τις δράσεις σε αυτό το τομέα. Θα δούμε να υπάρχει κάποια κάλυψη κατά πάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2010. Για τα κύρια θέματα κατά πάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το τέλη του 2010. Θέλω να σας τονίσω ότι η κατάσταση 2008-2009 ήταν ιδιάζουσα γιατί καταρχήν τέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, υπάρχουν νέες θέσεις που έχουν καθοριστεί. Και μετά που τέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα πια ένα άλλο καθεστώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νομικό καθεστώς με σημαντικές επιπτώσεις. Επίση, η, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγγνώμη, είναι υποχρεωτική τώρα. Και θα εφαρμόζεται και στο μέλλον. Και πάλι θα πρέπει να είμαστε καλύτερα ενημερισμένοι βέβαια στην πολιτική μας. Η οικονομική κρίση ανά τον κόσμο έχει επίση σημαντικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί όσον αφορά για το πληθυσμό που υποφέρει περισσότερο και αυτό καλύπτει από την έκθεση. Κλιματολογικέ αλλαγέ έχει επίση σημαντικέ επιπτώσει μακροπρόθεσμα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο ιδιαίτερα. Και επίση, μια σημαντική επίπτωση προέρχεται από τι σύγχρονε τεχνολογίε γιατί και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει μία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραδείγματος χάνω όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου. Αυτά γενικά, τώρα ορισμένε παρατηρήσεις στη δομή της έκθεσης. Έχουμε τα διάφορα κεφάλαια που καλύπτουν η έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. τα... Έχουμε τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνής Οργανισμούς, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κάθε γραμμή γραμμής Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανθρώπινα δικαιώματα ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και πολλά υποκεφάλαια θα μπορούσαμε να πούμε που αφορούν την δανειτική ποινή, την βία κατά των γυναικών, διεθνής ανθρωπιστικός, νο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και διάφορα άλλα που προέρχονται παραδείγματο χάρη από το Διεθνές Δικαστήριο. <clears throat> Όπως αναφέρθηκε, έχουμε 423 τροπολογίες, πάρα πολλές, και αυτό καταδεικνύει όμως πόσο σημαντική είναι η έκθεση, πόσο σημαντικό είναι το θέμα για μας. Ε, εγώ προσπάθησα να καλύψω όλες τις καταπληκτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλες τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τις δικές μου και τις πολιτικές μου ομάδες, αλλά όχι μόνον. Υπάρχουν 42 συμβαστικές τροπολογίες και θα ψηφίσουμε βέβαια υπέρ αυτών των συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλε τι οργανώσει προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου, που συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά μαζί μας. Ευχαριστώ για τι παρατηρήσει του. Το είπα και δεν μπορώ να, να επαναλάβω ότι οι προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικέ μη κυβερνικές οργανώσει είναι οι κύριοι μα σύμβουλοι και του ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή τους. Έχετε λάβει τις συμβαστικές απολογίες βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να τις αναφέρω μία προς μία. Απλώς θα ήμουν ευγνώμων στους συναδέλφους που θα συμβάλλουν τώρα στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ο κύριος Χόουιτ, πρώτος και ηγητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντρικίνα για την εργασία σας ως χήτρια εδώ σήμερα. Είχε αντιμετωπίσει ένα τεράστιο αριθμό τροπολογιών και να τις εξετάσει, να δει πού υπάρχουν επικαλύψεις, ποιες δεν είναι αποδεκτές κλπ. λοιπά και αναγκάστηκε να εργαστεί πολύ σκληρά για τις συμβαστικές προτάσεις και τις συγχαίρω εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για τη συνεργασία της ε, μαζί μας. και καμιά φορά μάλιστα στην Υποτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων δεν είχε πρόσβαση στην τροπολογία στη γλώσσα τη, παρόλα αυτά συνέχισε την εργασία, γιατί υπάρχει πίεση χρόνου. Εργάστηκε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα επίση να σα πω ότι θεωρώ ότι έχει σαγάγει κάποιε καινοτομίε αυτή την έκθεση. Παραδείγματο όσον αφορά την ελευθερία έκφραση στο διαδίκτυο. Η αναφερόμενοι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στον αφορά τη βία κατά παιδιών και γυναικών. Αυτή είναι μια ειδική συμβολή που έχει προσφέρει στην ε, ετήσια έκθεση. Και επίσης ε, αναφέρεται αναλυτικά στις εργασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, μια σημαντική συμβολή στην έκθεση φέτος. Είναι σημαντικό νομίζω η Άφετ να πει ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθήσαμε αυτή η έκθεση να μην είναι μια επικάλυψη ε, ή μια ελεκτική στην ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά προσπαθούμε να ελέγξουμε ακριβώς τις δράσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και των υπάτων εκπροσώπων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι πολύ καλό που βλέπουμε αυτή την, την προσέγγιση, γιατί βλέπουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πολλά σχόλια έχουμε για συγκεκριμένες χώρες, για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά είναι θέματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγουμε από την αναγκαιότητα της ε, προσέγγισης. Ε, ε, θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς θα μπορούμε κατά να είμαστε πολιτικά αποτελεσματικοί. Μία από τις τροπολογίες που υποβάλαμε εμείς ήταν να επιστήσουμε την προσοχή της υπάτου εκπροσώπου και του Συμβουλίου στο γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε μεγαλύτερη συμβολή του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία της έκθεσης κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, αν δεν κάνω λάθος. Ε, Είχαν πέσει ένα πιο δραστήριο ρόλο όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θέλαμε να επιθυμίσουμε στα άλλα θεσμικά όργανα ότι ακριβώς αυτό το να μιλάμε δηλαδή με μία φωνή είναι κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι καλύτερη προσέγγιση. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε δύο από τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, κύριε Αντρική, η μία όσον αφορά την έκθεση Goldstein, που ήταν δύσκολο να διαπραγματευτούμε ένα τμήμα της πρώτης αυτής. Υπήρχε μια συνέντευξη μεταξύ των μεγάλων πολιτικών ομάδων και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην ανοίξουμε τη δέσμη αυτής συμφωνίας και νομίζω ότι η κυρία Αντρίκεν ναι, πολύ επιτίδια βρήκε ένα συμβιβασμό κατάλληλο. Την ευχαριστώ γι' αυτό. Επίσης όσον αφορά το GSP+, υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις όσον αφορά πόσο αποτελεσματική και δίκαιη είναι η δράση της GSP. Και βρήκε και εκεί μια πάρα πολύ καλή τροπολογία η κυρία Αντρίκεν γι' αυτό. Όσον αφορά τις ε, σοσιαλιστικές προτεραιότητες, έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και λογικός ο συμβασμός που πετύχαμε όσον αφορά τους ομοφιλόφιλους. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά τις θρησκείες και τα πιστεύω, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια διάκριση κατά πόσον είμαστε κατά των διακρίσεων ε, της θρησκείας και βάσει των πιστεύω. Είναι μια σημαντική διαφορά αυτή. Ε, Επίση θέλω να πω ότι είναι πάρα σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίθετη με την ποινή. Όσον αφορά και τη φίλη κυρία Γκόμες, έχω να πω ότι έχουμε δύο κυρίες ιδέες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και τις Ευρωπαϊκές ε, Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κοινωνικές, ε, Οικονομικές και Πολιτιστικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλουμε να τα στηρίζουμε. Για τον Κουαντάναμο έχω να πω ότι ίσως αλλάξει η κατάσταση λόγω των δράσεων των ΙΠΑ τώρα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξουμε ιδιαίτερα σημαντικό, να αποδώσουμε ιδιαίτερα σημασία στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό. Και επίσης Θέλουμε να κάνουμε μια τροπολογία για να αναφερθούμε σε δύο χώρες που όχι πριν, αλλά τώρα ασχολούνται με την επανεγκατάσταση ε, κρατουμένων από το Γκοντάναμο. Καμιά φορά η δράση κάποιων κρατών μελών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δεν είναι πάρα πολύ αυτή που θα θέλαμε. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε πάντα να πετύχουμε ένα συμβασμό. Δεν είναι επικρίση αυτή η κατεξηγητή αλλά πραγματικά βλέπει ότι μεταξύ των πολιτικών μας ομάδων υπήρχαν πολύ μεγάλες αποχές απόψεων. Και είναι λυπηρό ότι η μόνη συμβαστική ε, τροπολογία που δεν μπορεί να στηρίξει η σοσιαλιστική ομάδα είναι η συμβασική τροπολογία 24 για την Κούβα. Γιατί πιστεύω όμως ότι μπορούμε να βρούμε ένα κείμενο που να καλύπτει όλους και ξανακάνω την προσφορά αυτή. Ίσως οι εμπειρογνώμονες το ΑΕΛΚΑ και οι εμπειρογνώμονες των σοσιαλιστών ακόμη και σήμερα το πρωί μπορούν να συνεργαστούν και να βρουν μια συμβαστική λύση και στον τομέα αυτών. Αλλά αυτό το είναι θέμα ε, από τα 500 που εξέτασε η εισηγήτρια δεν πρέπει να μας κάνει να μην ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία της κυρίας Αντρίκενε. Ο δεύτερος και ο εισηγητής, ο κύριος Ντόντσης. Thank you, Mr. President. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις τροπολογίες και για τους συμβασμούς. Χάρη στη συνεισφορά των συναδέλφων, η έκθεση πιστεύω στέλνει το σωστό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο προς τις τρίτες χώρες, τις συνεργασμένες χώρες, αλλά και προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν, κρατη και την ε, εξωτερική μας υπηρεσία. Δεν θα διστάσουμε να υπερψηφίσουμε λοιπόν γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για καλύτερο συντονισμό όλων των μηχανισμών και οργάνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, ως ε, σκιώδης για την ομάδα ALDE, θέλω να πω ότι θα υποστηρίξουμε τι περισσότερε τροπολογίες, όμω δεν πρέπει να περιληφθούν όλες στην τελική έκθεση. Θέλω να σημειώσω ότι η ομάδα μου θα καταψηφίσει ορισμένες τροπολογίες, όχι επειδή επί τη ουσία ε, διαφωνούμε, αλλά επειδή περιλαμβάνουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες ε, σε ένα τα άλλα εξαιρετικά ισορροπημένο κείμενο. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητε. Δεν μπορούμε ειδικά να αναφερθούμε σε κάθε ιδέα ή γεγονός όσο και αν αξίζει. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά εν κατακλείδη να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να σας καλέσω όλους να υπερψηφίσετε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουταλα είναι η τρίτη σκιώδης εισηγήτρια. Πρόεδρε, η προσθεμένη αξία αυτής της έκθεσης που θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο είναι ότι από τη μια γενική επισκόπηση της στρατηγικής μας όπως προσχέθηκε είπατε εκπρόσωπος. Είναι κάτι το οποίο περιμένει και η Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι πιστεύω ότι ως επισκόπηση της στρατηγικής μας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου το κείμενο πρέπει να είναι ανοιχτό, διαφανές, ε, ισορροπημένο. Θέλουμε, συνεπώς, να σε και μια ανακοίνωση ενδεχομένως της ε, Κομισιόν για να διευρυνθεί ο διάλογος σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική για τα δικαιώματα του ανθρώπου βάσει και της εθνικής της Λισαβόνας. Η κυρία Αντρική είναι κατά την άποψή μου, έκανε εξαιρετική δουλειά. Σύμφωνα με τις τροπολογίες, η εισηγήτρια ήταν εξαιρετικά ανοιχτή και σε άλλες προτάσεις που υπέβαλαν συνάδελφοι. Πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καλό. Ο κύριος Σούλτς από τους Πράσινους. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ε, ογκώδη και σοβαρή έκθεση που αναφέρεται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' αυτά πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις και συμπληρώσεις. Δεν θα πρέπει να αφαιθούμε μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά γενικά στα αναγνωρισμένα δικαιώματα του πολίτου, παραδείγματο χάρη το και παθητικό δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Και σε πολλές χώρες δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν αυτές οι νοθείες ε, της, ε, των εκλογών που βλέπουμε σε πολλά μέρη από τη Ρωσία μέχρι την Ουκρανία, το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Από την άλλη μεριά, αυτή η έκθεση θα πρέπει να διευκρινιστεί, παραδείγματο χάρη όσον αφορά τις επιθέσεις κατά των ε, δημοσιογράφων, όχι μόνο η περίπτωση Νατάλια στη Μυροβά, αλλά φέτος ε, σκοτώθηκαν 8 δημοσιογράφοι και 40 ε, εκπρόσωποι των ΜΜΕ έδειξαν πολύ κακών επιθέσεων. Ο Ρόμπερτ Κάσιν ήταν το τελευταίο παράδειγμα και αυτό θα πρέπει ίσως κάπου να το αναφέρουμε. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε τώρα πιο επίκαιροι. παραδείγματος χάρη έχουμε την περίπτωση των διαδηλώσεων για το άρθρο 31 του ε, Ρωσικού Συντάγματος. Είναι πολύ καλό που την περασμένη Κυρική πρώτη φορά ενεκρίθη μια τέτοια διαδήλωση. Συμμετείχα και εγώ, αλλά βέβαια ακόμα αυτό δεν είναι σύμφωνα με αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε όταν λέμε ελευθερία διαδήλωσης. Δηλαδή όταν επιτρέπεται μια διαδήλωση περιορίζονται όμως σε 800 συμμετέχοντας και υπάρχει στρατιωτική παρουσία της αστυνομίας ε, γύρω από τους διαδηλωτές αυτούς, δεν είναι καθαρή διαδήλωση όπως την καταλαβαίνουμε εμείς στις χώρες μας. Και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Γέγγελ, τελευταία τοποθέτηση. Η κυρία Γέγγελ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Αντρίκενε και όλους τους κοιόδους εισηγήτες. Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είδα πόσο έντονα ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Είδα τις πολλές τροπολογίες και εγώ συνεισφερά στις ε, προ... τροπολογίες αυτές και διαβάζοντας τώρα στις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, βλέπουμε ότι βέβαια δεν λύνονται όλα τα προβλήματα του κόσμου με την έκθεση αυτή. Αυτή η έκθεση όμως μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας στη νέα κατάσταση που βρισκόμαστε έχει ένα ειδικό βάρος. Αναφέρονται τα πιο σημαντικά θέματα για τις ε, χρονιές στις οποίες αναφέρεται η έκθεση αυτή. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το πλαίσιο που έχουμε και το έκανε πολύ καλά αυτό η συγγετρία. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσουμε ευρέως να τύχει ευρεία υποστήριξη η έκθεση αυτή γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να δείξει το βάρος του το κοινοβούλιο και να, αποτι... και να δούμε την έκθεση αυτή σαν μια βάση για μελλοντική εργασία και είδαμε πόσο εργάστηκε η συγκίτρια και την ευχαριστώ και την συγχαίρω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, η συγκίτρια έχει να κάνει κάποια συμπεράσματα. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στην συζήτηση για τις παρατηρήσεις τους τις προτάσεις και τις κρίσεις τους. Πριν περάσουμε στην ψηφορία, θα έλεγα για την Κούβα να συζητήσουμε περαιτέρω, να βρούμε μια σημαντική λύση. Δεν έχω αντίρρηση την για του συναδέλφου, αλλά θα ήθελα να κρατήσω το εφισταμένο κείμενο. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτού. DSP Plus ε, τα προβλήματα στο Γουαντάναμο Εκεί δεν έχω αντιρρήσει. Ευχαριστώ και για τον σκιώδη εισηγητή από την Άλτε Ο κ. Σούλτς ανέφερε τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις παραβιάσεις του στην Ρωσία. Έχει απολύτως δίκιο. Δεν είναι Ιταλία μόνο, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι βρήκαν το θάνατο πρόσφατα στην Ρωσία. Ακούσαμε και για άλλες περιπτώσεις και παρακολουθούμε τις διαδηλώσεις στη Ρωσία. Βλέπουμε πώς τις αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι. Η κατάσταση θεωρώ ότι κατά τη βελτιώνεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλάμε για την περίοδο 2008-2009. Άρα αυτό πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο μα, Φυσικά θα λάβουμε υπόψη μα και τι εξελίξει το 2010, αλλά η περίοδο αναφορά, επαναλαμβάνω, είναι 8 και 9. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε και στο 2010, εννοείται. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω λοιπόν στην ε, ψηφορία μα με το απόγευμα. E λοιπόν, σας θυμίζω ότι θα ψηφίσουμε το απόγευμα. Και θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου με την ύπατο εκπρόσωπο την κυρία Άστον. Τώρα, επόμενο σημείο. 5. Βιώσιμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απότερο βορρά, αλλά δεν είναι παρόν ο εισηγητής. Διακοπή λοιπόν πέντε λεπτά. Bene, possiamo riprendere. Ξαναρχίζουμε. Το σημείο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η βιώσιμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απότερο βοριά. Μετά από την ακρόαση που είχαμε στις 2 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Γκάλερ ετοίμασε ένα πρώτο κείμενο το οποίο θα συζητήσουμε. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, κύριε Γκάλεχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τον να ασχολείται κανείς με τον απότερο βορρά και την ε, εξέλιξή του και ανάπτυξή του είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πόσοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, ποιοι είναι οι προγραμματιστές, πόσες συμφωνίες ισχύουν, ποια είναι τα νομικά καθεστώτα που ισχύουν σε αυτή την περιοχή. Και προσπαθώ να δω από πού ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 και πώς μπορεί να δράσει ούτως ώστε να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της εργασίας μας θα πρέπει να είναι να υιοθετήσουμε μια έκθεση που να λαμβάνει υπόψη την τροποποιημένη γεωπολιτική κατάσταση γύρω από την Αρκτική. Και όλοι οι ενδιαφέρομενοι να ξέρουν ακριβώς ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς σκέφτεται να δεσμευτεί η Ευρώπη στην Αρκτική. Ακόμα και αν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παράλληλα στην Αρκτική, με την Γρυλανδία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εξαρτάται από την Δανία, Φιλανδία, Σουηδία εκπροσωπούμεθα στην ευρύτερο χώρο της ε, αρκτικής ε, περιφέρειας και με την υποψήφια χώρα Ισλανδία επίσης. Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και υπάρχουν και άλλες εταιρικέ σχέσεις που αναφέρονται και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχουν, ε, μαζεύονται μάλλον τα κατάλοιπα της μόλυνσης της ε, ατμόσφαιρας και των υδάτων και γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα. Στην προσημασία της έκθεσης, εκ μιας αρχής συνεννοήθηκα με τους σκιώδες συζητητές, είχαμε διάφορες συναντήσεις και μίλησα και με ορισμένους από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Καταρχήν προσπάθησα στην έκθεση να αναπτύξω τους τομείς πολιτικής που παίζουν σημαντικό ρόλο στα σημεία 1 3 και είπα ότι ορισμένε από τις πολιτικές αυτές είναι και θέματα της κοινότητας και αναφέρθηκα εκ μιας αρχής σε εκείνους που κατοικούν στην ε, ακτική περιοχή, γιατί για αυτούς εργαζόμαστε. Περιβάλλον, πολιτική για το κλίμα, έρευνα, ε, ναυσιπλοεία, αλία, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Προσπάθησα να αναφερθώ στο θέμα των προτεραιοτήτων των άμεσα εγκαταστημένων εκεί και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα συνεργασίας. Στόχος της έκθεσης είναι να τονίσουμε πώς θα είναι πιο συμβατά τα διαφορετικά συμφέροντα. Ακριβώς επειδή γεωγραφικά δεν είμαστε ακόμα κάτοικοι των οχθών εκεί της Αρκτικής θάλασσας. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό θα το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει ακριβώς όπως είπα να προωθήσουμε μια ανηφόρα ανάπτυξη και με την περιοχή αλλά και με τους κατοίκους, τους πολίτες που ζουν εκεί. Όσον αφορά ε, το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος, αλληλεία και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στους τομείς αυτούς θα πρέπει στο υψηλότερο δυνατό τεχνικό επίπεδο να φροντίσουμε, να αναφερθούμε όχι μόνο στις στόχους, αλλά στην πράξη. Και γι' αυτό λέω ότι μέσα στα πλαίσια της ΕΜΟ, της Διεθνούς ε, Οργάνωσης για τη Θάλασσα και μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου της Αρκτικής επίσης, να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Αναφέρω επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τον έλεγχο του 40% του διεθνούς εμπορικού στόλου. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο λόγω των αλλαγών των κλιματολογικών πολιτικά θα πρέπει να εξελευθούν επίση διαφωνίε που υπάρχουν παραδείγματο χάρη μεταξύ Νορβηγία και Ρωσίας. Μια που εμεί είμαστε καταναλωτέ των πόρων αυτών, Όπω το προανέφερα, έχουμε κάθε συμφέρον για συνεργασία, ιδίω όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα. Και αυτό γίνεται κυρίως με τεχνολογικές μεταφορές που θα πρέπει να είναι δυνατές προς όφελος και των με και των δε. Η μεταφορά αυτή του υψηλού κατά του επίπεδου τεχνολογίας είναι σημαντική γιατί έχουμε το 1 πέμπτο περίπου στην περιοχή αυτή των γνωστών αποθεμάτων ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων φυσικών πόρων. Αυτή η αηφόρος κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει η Αρκτική να ανοίξει και να το θεωρήσουμε αυτό σε μια ευκαιρία, όχι μια απειλή να προασπίσουμε τα συμβαίνοντα των πληθυσμών και των ηθαγενών πληθυσμών που θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη. Εγώ συζήτησα με μία εκπρόσωπη των που μας είπε ότι δεν θέλω να ζω σε μουσείο τελικά, δηλαδή στην ανάπτυξη της Αρκτικής δεν πρέπει να, προσ... να προσπίσουμε τα σφαίρα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα φυσικό πάρκο, αλλά να υπάρχει μια αηφόρος ανάπτυξη στην περιοχή αυτή το θέμα της σωστής διακυβέρνησης. Αναφέρθηκα ήδη στους ε, κανόνες και θεσμικά όργανα που υπάρχουν και στο Ακτικό Συμβούλιο και καλό το Συμβούλιο αυτό να είναι πιο ενεργό και να ε, υιοθετεί και κανόνες δεσμευτικούς. και ότι θα ήταν καλό ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλουμε ένα μόνιμο εκπρόσωπο στο Συμβούλιο αυτό. Αυτή τη στιγμή ε, εκπροσωπούνται τα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά θα ήταν καλό και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπείται <clears throat> και νομίζω και πριν από τις συνθήκες Λισαβόνας είχαμε πολλές αρμοδιότητες κοινοτικού τύπου. Και θα πρέπει και εδώ νομίζω να έχουμε μία μόνιμη εκπροσώπηση. τα τελικά συμπεράσματα στο οποίο καταλήγω με την έκθεσή μου είναι αφενός στα πλαίσια της Γενικής ΜΑΡΕ στην Κομισιό να υπάρχει μία μόνιμη δομή υπηρεσιών που να επιτρέπει μία συνεπή εργασία, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά τους ερευνητικούς πόρους όχι μόνο για την Αρκτική, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω το σύνολο της ε, περιοχής της Αρκτικής θα πρέπει να ωφελείται από ειδικά ταμεία χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότηση, ώστε μπορέσουμε έτσι αποτελεσματικά να δράσουν στον τομέα της έρευνας. Εγώ είμαι υπέρ ενός αρκτικού κέντρου ενημέρωσης σαν ένα μέσο της κοινωτικής πολιτικής για να ενημερώνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στην Αρκτική για τη δική μας πολιτική και από την άλλη μερία να συλλέγουμε πολιτικές ε, δικές τους. Προτείνω επίσης το πρόγραμμα Γαλιλαίο και άλλα δορυφερικά προγράμματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε να χάρη την ασφάλεια των θαλασσών και θεωρώ ότι τα μηνύματα που αποστέλουμε όσον αφορά τη δέσμευσή μας Αυξάνουμε το δυναμικό κοινή συνεργασίας και μπορούμε έτσι να πετύχουμε υψηλά πρότυπα στην προστασία των θαλασσών. Και εν κατακλείδη έχω να σας πω ότι ακριβώς άμα ασχοληθεί κανένας με το θέμα αυτό, αποκτά τόσες πολλές ιδέες και προτάσει που δεν μπορούσα εγώ να εκμεταλλευτώ εδώ στην έκθεση γιατί είναι πολύ περιορισμένη. Εξαρτάμε λοιπόν και από το αυτό θα μπορούσα να προτείνουν σαν τροπολογία οι σκιώδες συζητητές. Ε, κατά τα άλλα έχω και εγώ κάποιες τροπολογίες που θα μπορούσα να προτείνω. Είναι αγκασμένος κανένας να εφαρμόζει αυτά τα διάφορα κόλπα εάν ο οι δυνατότητε που έχει μέσα στη συνέχιση αυτή καθ' αυτή είναι περιορισμένε. Ευχαριστώ όλου του συνέβαλαν μέχρι στιγμή και ευχαριστώ και εκείνου που θα συμβάλλουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Γκάλερ. Η κυρία Γιάκονσάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλε. Πρόκειται για ένα κείμενο Πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο συνάδελφος Γκάλερ το έχει εξετάσει εις βάθος το θέμα. Τον ενδιαφέρει λοιπόν. Τώρα, για αυτήν την ανάλυση, μία κριτική για να ξεκινήσουμε. Σε αυτή την έκθεση διαπιστώνουμε ότι η Αρκτική ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο και αυτό εξαιτίας των ε, κλιματικών αλλαγών αποτελεί και θεωρούν πολλοί ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που καθιστά επίκεντρο προσοχή στην Αρκτική. Εγώ θεωρώ το αντίθετο <clears throat> όμως. Θεωρώ ότι είναι οικονομικές προκλήσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον για την Αρκτική. Υπάρχουν τεράστιοι φυσικοί πόροι εκεί και όλοι θέλουν να τους εκμεταλλευτούν. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε Πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν τι είναι κλιματική αλλαγή και τι είναι το οικονομικό ενδιαφέρον, διότι τελικά μπορούμε να έχουμε από την Αρκτική την κάλυψη του ενός τετάρτου των ε, ενεργειακών μας αναγκών. Ή, βέβαια τα νέα δεν είναι μόνο κακά, έχουμε και καλά νέα. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις, η ανάπτυξη στην Αφρική πάντα εκτυλίχθηκε ειρηνικά. Είδατε τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και καλα νεα βλεπουμε οτι η εξελιξεις η αναπτυξη στην αφρικη παντα εκτιλήχθηκε ειρηνικα ειδατε τη συμφωνια μεταξυ ρωσιας και νορβηγιας για τον έλεγχο των συνόρων, για τον έλεγχο του πετρελαίου. Έχει λυθεί λοιπόν όλη αυτή η υπόθεση. Βλέπουμε ότι όλα τα εξελίσσονται ειρηνικά. Γιατί διότι στην Αρκτική έχουμε μια μεγάλη παράδοση διασυνοριακής συνεργασίες. Επίσης υπάρχει μια γενική, ένα γενικό πνεύμα που βλέπει τους πληθυσμούς εκεί. Υπάρχει η φυλή των Σάμις οι οποίοι ε, θεωρούν τον εαυτό τους πολίτες του κόσμου και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για σύνορα. Εμείς λοιπόν δεν βρισκόμαστε εκεί για θέματα εξουσίας, όχι. Βρισκόμαστε εκεί για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν θέλει να διεισδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή και ο Καναδάς εξάλλου δεν το θέλει πολύ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λύσουμε το πρόβλημα. Διαπιστώνεται επίσης ότι το Συμβούλιο της Αρκτικής θα πρέπει να ενισχυθεί, διότι σε αυτή τη φάση είναι, αποτελεί μάλλον το μόνο λαϊκό βήμα, το μόνο λαϊκό φόρουμ όπου συνεργάζονται όλοι και συμμετέχουν και οι ηθαγενείς. Βέβαια το όργανο αυτό δεν είναι ακόμη ενισχυμένο, δεν έχει γραμματεία, δεν έχει μία δομή, δεν έχει οργάνωση. Ξέρω ότι η κυρία Άστον έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα γύρω από αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο της Αρκτικής είναι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παλέψει περισσότερο για να ενισχύσει τις σχέσεις με, με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τη Ρωσία για την περιοχή, για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη θα πρέπει να δημιουργήσουμε δίκτυα, ε, δί, ε, δίκτυα έρευνας, αναπτυξιακά δίκτυα, χρηματοδότηση κοινή για την έρευνα. Γίνεται έρευνα στην Ιταλία, στην Ορβηγία, στη Φιλανδία, παντού. Αλλά λείπει συντονισμό. Θα ήθελα σε αυτή την έκθεση να τονιστεί ο ρόλος της βόρειας διάστασης, αυτό το παράθυρο στην Αρκτική διότι υπάρχει το δίκτυο συνεργασίας με τη Ρωσία που είναι και το μεγαλύτερο σήμερα στην Ευρώπη δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στις τηλεοράσεις αλλά είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τη Ρωσία σε αυτό το παράθυρο της Αρκτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να παίξει έναν αρχηγικό ρόλο και για την οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε τις βάσεις και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο συνάδελφος Γκάλερ μίλησε για αυτό το κέντρο κατάρτισης, συγγνώμη, κέντρο έρευνας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας για την Αρκτική. Είναι πολύ ωραία ιδέα διότι χρειαζόμαστε στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία. Χρειάζεται μία πολυκλαδική επιστημονική εστίαση. Και αυτό το κέντρο θα μπορούσε να έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας. που είναι και η βάση της, ε, του Αρκτικού Πανεπιστημίου. Μιλάμε λοιπόν για τους αυτόχθονες, αλλά δεν μιλάμε για τους ντόπιου. Αυτό είναι λάθος. για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών. Δεν θα πρέπει να μιλάμε λοιπόν μόνο για τους αυτόχθονες, αλλά για όλους τους κατοίκους. Επίσης, δεν αναφέρεται καθόλου και η οικονομία του τάρανδου. Μιλάμε για πετρέλαιο, για άλλα πράγματα, αλλά δεν μιλάμε για τους ταράνδους. Η τάρανδη για τους ντόπιου είναι σημαντικό έσοδο. Η ελία το κυνήγι, πολύ πολύ πιο σημαντικά για τους ντόπιου από ότι προμήθεια σε φυσικό αέριο. Για να μπορέσουμε λοιπόν εμείς να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, σχέση εμπιστοσύνη με τους ντόπιου. Πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις δραστηριότητές τους, διότι οι αυτόχθονες ε, σοκαρίστηκαν πάρα πολύ από τις αποφάσεις που είχαμε σχετικά με το κυνήγι της Φώκιας κλπ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερ εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας. Έχουμε ένα λοιπόν σημαντικό έγγραφο οποίο προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Η κυρία Γιάτεν Μάτ. Πρόεδρε, τα φιλανδικά ονόματα όντω είναι ε, καμιά φορά δύσκολα. Εσείς όμως ε, μια χαρά τα πείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλερ για την έκθεση που συνέταξε. Πρόκειται για το πρώτο σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αποδερό Βορρά. Ιστορική λοιπόν η στιγμή. Άλλωστε ήταν καιρός να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για τη διάθεση συνεργασία που έδειξε με του κοιόδη συγητέ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένη από την έκθεση του κύριου Γκάλερ. Έχει εξαιρετικά στοιχεία. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διάσταση της πολιτικής για τον απότερο βορρά. Θα έλεγα ότι η πολιτική για τον απότερο βορρά πρέπει να αποτελέσει τη της υφιστάμενης πολιτικής για τον βορρά εν γέννη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη τέτοια πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι η αρκτική πολιτική, πολιτική για την αρκτική πρέπει να επεκταθεί, να ενισχυθεί ως μέρος ενός συνόλου και όχι αποσπασματικά και ξεχωριστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ή άλλως στην Αρκτική, έχει συνεργασίες στον τομέα, για παράδειγμα, της πυρηνικής συνεργασίας, την διαχείριση των λιμάτων, την περιβαλλοντική προστασία και κοινωνικά μέτρα. Φυσικά υπάρχει πεδίο για περαιτέρω συνεργασία. Η βόρεια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεράζει τις χώρες της ε, Αρκτικής, μεταξύ άλλων την Ρωσία, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Πρόκειται για σημαντικούς εταίρους στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βόρεια διάσταση. Και φυσικά έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά με τους οποίους συνεργαζόμαστε, διότι είναι παρατηρητές στο πλαίσιο αυτό. Το δεύτερο σημείο αφορά το κέντρο πληροφόρηση για την Αρκτική. Θεωρώ ότι το σχετικό δίκτυο πληροφόρησης πρέπει να το αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα. Όπως είπα σε αυτήν την Επιτροπή αλλά και σε άλλα φόρα. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα για να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που τεκταίνονται αυτήν την στιγμή στην Αρκτική, τόσο αφορά το κλίμα αλλά και άλλους τομείς. Πέρα από τα ευρωπαϊκά όργανα, το δίκτυο και το κέντρο πληροφόρησης της Αρκτικής, πρέπει να φροντίσουμε να υπηρετούν το κοινό καλό και την κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, όπως η Λίσσα Γιάκονσάρη είπε, η αδελφός μου, θα έβλεπα με καλομάρι το κέντρο να έχει την έδρα του σε πρώτη βόρεια περιοχή, μαζί ίσως με το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας. Εκεί έχουν ένα ερευνητικό κέντρο και έχουν κάνει πολλά για τα σχετικά θέματα. Το τρίτο σχολείο μου έχει σχέση με το εξή. Και εγώ θέλω να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να τους αγνοούμε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική. Οι σαμογέτες έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ανοιχτό διάλογο με τους σαμογέτες. Συνεπώς, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην ανακοίνωση της Επιτροπής το 2008 για την Αρκτική γίνεται ρητή μνήα αυτής της ανάγκης. Ας το κάνουμε λοιπόν, όπως ούτως ή άλλως η Κομισιόν πρότεινε να γίνει. Διάλογος λοιπόν με τους ομογέτες. Και επιπλέον, οι ομογέτες της Φινλανδίας και της Σουηδίας δεν έχουν μόνιμη εκπροσώπηση αποστολή τη Βρυξέλλε. Συνεπώ η φωνή του δεν ακούγεται στην πράξη. Αυτά είναι τα τρία σχολιά μου. Δίκαιο μεταυτοχθόνων, βορειοδιάσταση και κέντρο πληροφόρηση για την Αρκτική. Αυτά πιστεύω ότι πρέπει να τονιστούν περαιτέρω. Κατά τα άλλα, η έκθεση είναι εξαιρετική. Κύριε Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. κυρία Λέζινγκ. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση και είδα ότι εσείς κύριε Γκάλερ μιλάτε για το περιβάλλον, για τη γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική, τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και μιλάτε και για ασφάλεια. Λείπει όμως κάτι κατά τη γνώμη μου. Και είναι ίσως σημαντικό για το μέλλον, είναι η διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των πτυχών και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έχουμε τη συνεχή ρήπανση της περιοχής, την αύξηση της ρήπανσης στην περιοχή και η βιομηχανική ανάπτυξη με την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και η διεύρυνση των συμπορικής αερίας και στην περιοχή αυτή οδηγεί σε παρεμβάσεις και μόλυνση του ευαίσθητου οικολογικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω στην έκθεση να υπάρχει μια πιστική στρατηγική εάν προχωρήσουμε έτσι όπως προβλέπετε. Πώς θα διορθωθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση. Αναρωτιέμαι κατά πόσον υπάρχουν και άλλες εξελίξεις και άλλες ιδέες, κατά πόσον η Κομισιόν έχει μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση. Το κύριο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, περιοχή της Ακτικής να δράσει είναι ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τήξη των ε, παγοβούνων εκεί όπως είπαμε υπάρχουν καινούριε ε, θαλάσσιοι οδείοδοι, υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν υπήρχε προηγουμένως γιατί ήταν κάτω από τα στρώματα πάγου και ακριβώς η στρατηγική κλίματος του Μαρτίου του 2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει αυτά τα σημεία. Δεν θέλω να τα επαναλάβω ένα προς ένα, αλλά και εκεί αναφέρεται η βελτίωση ε, η βελτιωμένη συγγνώμη πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και το θέμα της ε, διεθνούς σταθερότητας και θέματα της ε, ασφάλειας. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα συζητήσει και αυτό οδηγεί και σε γεωστρατηγική σημασία της Αρκτικής. Η Ρωσία οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Νορβηγία, η Δανία, ο Καναδάς ξεκίνησαν μία στρατικοποίηση της Αρκτικής. Το 1999 ο Αμερικανικός στρατός ξεκίνησε την εφαρμογή της roadmap για την Αρκτική, του δικού χάρτη για την Αρκτική. Χρειάζεται λοιπόν σκέψη γύρω από όλα αυτά. Για το αν θα πρέπει να έχουμε συνεχώς στρατεύματα στην Αρκτική, δηλαδή μόνιμες στρατιωτικής βάσης. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με την Αμερική, αλλά και ο Καναδάς ξεκινάει σχέδια. Και η Ρωσία είπε ότι το 2020 και μετά θα δημιουργήσει μια ειδική δύναμη, στρατιωτική δύναμη για την Αρκτική για να μπορέσει να περιφρουρεί τα στρατηγικά της συμφέροντα στην περιοχή. Αλλά μου λείπει Μου λείπει σε αυτήν την έκθεση μία, ανάλυση για, την... για τις ε, περιβαλλοντικές αλλαγές. Η Αρκτική δεν μπορεί να αποτελέσει, να αποτελέσει στο μέλλον μία νέα λεκάνη κρίσεων. Χρειάζεται να έχουμε μία μετριοπαθή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Αρκτικής, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τις προάλλες εγώ είχα μιλήσει για μια συνθήκη για την Αρκτική, αλλά μου το κόψανε αμέσως, μου είπανε ότι δεν έχω δίκιο και ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτιέμαι... Δεν ξέρω, δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια σύμβαση ή δεν υπάρχει βούληση για τέτοια σύμβαση, γιατί το περιεχόμενο συνθήκης αυτή θα πρέπει να είναι ένα μορατόριουμ για την εξόριξη των φυσικών ε, πόρων από την περιοχή χ εκείνη. Αυτό που αναφέρθηκε συχνά εδώ ήταν το θέμα των αυτοχθόνων και θα ήθελα να το διευκρινίσω και να αναφερθώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες περιοχές ε, του κόσμου. Πού αλλού υπάρχει ε, η παρουσία τόσων πολλών χωρών που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους στις περιοχές αυτές και πού οδήγησε τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε αυτές τις άλλες περιοχές. Και όταν συζητάει κανένας με κάποιον, ε, δεν πρέπει να συζητάει με αυτούς που ίσως θα εκμεταλλευτούν, θα ωφεληθούν από την εξέλιξη αυτή. Να μιλήσει κανένας με τους χωρικούς, ε, με όλες τις ε, πτυχές, όλα τα στρώματα του πληθυσμού που θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και που φοβούμε ότι μακροπρόθεσμα θα έχουν αρνητικέ επιπτώσεις από την εξέλιξη αυτή. Ευχαριστώ. Bene, la parola all'ultimo relatore a ombra, l'onorevole Tarant. Oh, κύριος Τάραντ που είναι ο τελευταίος και ο εισηγητής. Έναν, herra president. Ja yeah. kui lubate, ma jätkan Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και εγώ μια γλώσσα της Αρκτική. Ε, Αρκτικής. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Γκάλα και να τονίσω ορισμένα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την ομάδα των Πρασίνων. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να στηρίξουμε την Αρκτική είναι μια διεθνής συνθήκη για το κλίμα, η οποία θα είναι δεσμευτική. Απουσία όμως τέτοιες ε, συνθήκες σας κάνουμε λιγότερα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες για τις ε, εκπομπές άνθρακα. Το ίδιο έχουν κάνει και τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε λοιπόν εδώ κάποια μέτρα. Ε, τώρα όσον αφορά την εξόριξη πετρελαίου και αερίου, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η τεχνολογία δεν έχει οριμάσει ακόμη για την εκμετάλλευση αυτών των πόρων στην περιοχή της Αρκτικής. Πιστεύω ότι η απληστία της ανθρωπότητας την σπρώχνει στην Αρκτική. Όπως είπε και η συνάδελφος ε, Λέζινγκ, οι συνθήκες μπορεί να είναι από γεωλικής απόψης διαφορετικές στο βορρά και στον νότο, αλλά το νομικό πλαίσιο πρέπει να, να είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προλάβει αυτή την καταστροφή στην Αρκτική. Τώρα για το Συμβούλιο της Αρκτικής. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε παρατηρητές. Η Νορβηγία δήλωσε ότι θα αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή και πιστεύω ότι και οι Φιλανδοί και άλλοι θα κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα έχουμε λόγο σύντομα στο Συμβουλίο της Αρκτικής. Το Συμβουλίο της Αρκτικής βεβαίως δεν έχει καν μόνιμη γραμματεία. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει ένα τέτοιο, άλλο ένα μάλλον, γραφειοκρατικό όργανο. Το κέντρο ερευνών τώρα στο Ροβανιέμι πρέπει να ειδηθεί εκεί, στο Ροβανιέμι, όχι στις Βρυξέλλες. Επίσης το θέμα του κυνηγιού της ε, φώκιας είναι ένα σημαντικό θέμα. Το σημερινό κείμενο πρέπει να ενημερωθεί διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μεταξύ, όπως ίσως γνωρίζετε, εξέδωσε απόφαση η οποία δεν συνάδει πλήρω με τους πολιτικούς μας τουλάχιστον στόχους. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν και δύο προτάσεις. Η μία για την ε, διεθνή ναυτιλία για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη και είναι μια πρόταση με την οποία συμφωνώ. Όσον αφορά τώρα την σύγκρουση Αμερικανών και Ρώσων δεν νομίζω να είναι πολύ πιθανή αλλά πρέπει να επικρατήσει σύνεση όσον αφορά την χρήση των φυσικών πόρων. Να αποφύγουμε ένα νέο κύμα άπλης εκμετάλλευσης στην Αρκτική. Επίσης, ε, αναφέρθηκε συνάδελφος ε, στα δικαιώματα των αυτοχθόνων και αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Οι οι οποίοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια έχουν φωνή στην αντίστοιχη πρωτεύουσά τους. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι παραπάνω σε διαστολή με αυτό που έχουν ή μάλλον δεν έχουν οι Καναδοί αυτόχθονες. Η ουσία βεβαίω είναι πιο σημαντική, αλλά εάν χρειαστεί και αυτή η μόνιμη αντιπροσωπεία, να την έχουμε. Νομίζω όμω ότι μίλησα πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, αυτά προς το παρόν. Έχουμε τρεις ακόμη μιλητές. Ο κύριος Σούλτς, ο Ταλαντσπέρκης και ο Τάλα. Σας παρακαλώ να είστε ακόμη πιο σύντομη, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θα ήθελα ρητά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τόσο μεγάλη του δέσμευση και αυτό ε, οδήγησε και σε μια μεγάλη ε, ακρόση που είχαμε εδώ, γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για ένα θέμα που δεν έχουμε ακόμα τονίσει επαρκές από την έκθεση ΣΥΠΡΕΣ του Ινστιτούτου Έρευνα Ειρήνη τη Στοκχόλμη, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και θα πρέπει πραγματικά να δούμε τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το καθεστώ του παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να αποφύγει μια σύγκρουση των μεγάλων δυνάμων δυνάμεων για τις ε, θαλάσσιες ε, διόδους ή για την εκμετάλλευση των η κυρία Λίζιν τα είπε όλα αυτά που είχα να πω. Θα μπορώ να είμαι σύντομος. Βλέπουμε να υπάρχει ε, στρατιωτική ε, ε στρατιωτικό εξοπλισμό και η Ρωσία μάλιστα τοποθετεί και μια σημαία στο βυθό τη θάλασσα για να δείξει πραγματικά τι απαιτήσει έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο Λαντσπέργη έχει το λόγο. Uh, you, Πρόεδρε, του κυρίου Μιχαήλ Γκάλερ όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί του Βορρά είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Ζούμε σε περιβάλλον εντάσεων. Δεν χρειαζόμαστε άλλες εντάσεις. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια σχετική δήλωση. Ο εισηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασία. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο διεθνής ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω εντάσεις. Εδώ υπάρχει ίσως ε, ένα μικρό μειονέκτημα του κειμένου. Θα πρότεινα λοιπόν στον κύριο Γκάλερ να τονίσει αυτή την πτυχή. Και ελπίζω να μην αργήσουμε να κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Επίσης, το εκτιμώντας H, το αγγλικό κείμενο, επιτρέψτε μου να κρατήσω μια τροπολογία, η οποία έχει ως εξής. Δεδομένου ότι ήδη εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε κινήσεις ε, χωρών να διεκδικήσουν χώρο ακόμα και τον βυθό. Θεωρούμε ότι πρέπει να προληφθεί ε, άλλη μία απεικιοκρατικού τύπου επέκταση στην περιοχή. Αυτήν την ανησυχία σχετικά λοιπόν με τις ε, κτηρικές διαθέσεις ορισμένων χωρών στην περιοχή, αυτήν πρέπει να την εκφράσουμε. Αουτάλα, τελευταία παρέμβαση. Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Ταράν και την κυρία Γετεμάκη για το γεγονό ότι θα μπορούσαμε να πούμε λίγο περισσότερα για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Θέλω να τονίσω ότι στην περιοχή, στην Αρκτική, ζουν πολύ μικροί λαοί. Πέρα από τους αυτόχθονες Χάνση και Μάνση που ζουν για παράδειγμα στα βόρεια της ε, Φιλανδίας. Η ανθρώπινη λοιπόν διάσταση πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Γιατί στι περιοχέ αυτές ζουν άνθρωποι και όχι μόνο οι αυτόχθονε, αλλά και άλλοι. Συνεπώ, ω Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσουμε για τις γλώσσες τους, τι οποίε έχουν δικαίωμα να περάσουν στα παιδιά του και τα εγγόνια του. Οι άνθρωποι λοιπόν που μιλούν τις τοπικές γλώσσες να μπορούν να συνεχίσουν να μιλούν τις γλώσσες τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλιώς αυτές οι γλώσσες βαίνουν προς εξαφάνιση. Στην εισαγωγή αναφέρονται διάφορες ε, συμβάσεις, συμφωνίες. Πιστεύω ότι τουλάχιστον τους Αμογέτες και τους Βόρειους Αμογέτες και τις σχετικές συμφωνίες, συμφωνίες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, αυτά θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε εκεί με έμφαση στα δικαιώματα στην γη και σε άλλες ε, δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν πως θέλει ο κύριος ο δόκτωρ Γκάρθης Τελοσφάγιος. Πρόεδρε, εκ μέρους της Κομισιόν θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την ε, πλήρη ικανοποίησή μας για την έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μας έχει μεγάλη σημασία να ακούμε απόψεις και ιδέες όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απότερο βορρά. Αυτό ικανοποιεί και την Κομισιόν και την Μελλοντική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχω λοιπόν στα χέρια μα σημαντικά στοιχεία για την χάραξη πολιτική. Να σχολιάσω όμως ορισμένα από τα ζητήματα που έθιξαν οι προλαλήσαντε. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι δεν έχουμε άμεσα σύνορα ή ενδιαφέροντα στην Αρκτική, δεν έχουμε σημαντική παρουσία γενικά στην Αρκτική, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε απόντες. Δεν ε, βλέπω γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι μέρος του παιχνιδιού στην Αρκτική. Μετά έχουμε και την προοπτική η Ισλανδία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φυσικά θα ανέτρεπε ριζικά την κατάσταση. Ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν σε αυτήν την ε, πολιτική για τον απότερο βορρά, στο πλαίσιο της βόρειας διάστασης. Αυτό το σχόλιο ήταν πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η βόρεια διάσταση είναι πλέον μια κοινή πολιτική μαζί με τη Ρωσία, την Ορβηγία και την Ισλανδία. Δεν είναι απλώς κοινωτική πολιτική. Η πολιτική που προτείνει λοιπόν η Κομισιόν το 2008 και την οποία έχει λάβει υπόψη του το Συμβούλιο, εδώ μάλιστα το Συμβούλιο και το Πράσινο Φως πρόσφατα, η πολιτική αυτή λοιπόν έλεγα είναι η αρκτική πολιτική, η πολιτική για την αρκτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν εμείς να αξιολογήσουμε πλήρως αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει και πρέπει να τονίσουμε ότι, και, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μια δύναμη της, της Αρκτικής και θα πρέπει να τονίσει το ρόλο της στην περιοχή. Συμφωνούμε επίσης στη σημασία του διαλόγου με τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε ότι δεν είχαμε διάλογο με την φυλή Σάμι. Είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι μόνοι οι αυτόχθονες ε, που <coughs> ε, πληθυσμοί που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν συζητήσαμε μόνο με τους Σάμι, συζητήσαμε και με άλλες φυλές της Αρκτικής και το Μάρτιο και σε άλλες μελλοντικές συνεδριάσεις θέλουμε να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα ενδιαφέροντος για όλους τους πληθυσμούς. Θέματα υγείας, θέματα παιδείας είναι πολύ σημαντικά για αυτούς. Και όπως είπε και μία βουλευτής προηγουμένως, έχουμε αυτόχθονες πληθυσμούς που μιλούν ε, μία διάλεκτο μεταξύ φιλανδικών και ουγγρικών και που ε, δεν ε, ε, έχουν ιδιαίτερες διευκολύνσεις στην Ρωσία. Ευχαριστούμε επίσης για το ότι γίνεται αναφορά στη δημιουργία υπηρεσιών ε, αρμοδίων για την Αρκτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σίγουρα υπάρχει η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ η οποία είναι μια εγκάρσια σε οργάνωση σε διεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να έχουμε και μια ειδική υπηρεσία. Μιλάμε για περιοχές ε, κυρίαρχων ε, κρατών ε, για πληθυσμούς που είναι ριζωμένοι εδώ και χιλιετίες στην Αρκτική και πρέπει να διαπραγματευτούμε με όλους αυτούς. Θυμίζω λοιπόν ότι 15 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι λήγει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αμάν ξέχασα, λέει ο Πρόεδρος, ξέχασα τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συναδελφοί για τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Οπωσδήποτε. Για τους λόγους που προανέφερα, θα λάβω υπόψη με ορισμένε από τα αυτό για τους αυτόχθονες πληθυσμούς δεν μπορούσα να το λάβω υπόψη μου στη σχέδιο της έκθεσης, γιατί δεν είχα αρκετό χώρο και είναι, είμαι ευγνώμη που θα υποβάλλεται μια τέτοια η συνάδελφος Αγωνσάρη είπε ότι οι πρώτες τροπολογίες ε, προέρχονται από την ε, βιομηχανία και όχι από τις ανάγκες ε, αντίδρασης στις κλιματολογικές αλλαγές. Εγώ θα θέλω να το θέσω επίσης όρις και στην αρχή. Η παγκοσμιοποίηση αλλά και οι κλιματολογικές αλλαγές μας υποχρεώνουν να ασχοληθούμε με την περιοχή αυτή. Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ μόνο στους αυτόχθονες πληθυσμούς, αλλά και στους τόπιους κατοίκους που ζουν εκεί χωρίς να είναι αυτόχθονες. Και σας είπα και ήδη οι αυτόχθονες λένε ότι δεν θέλουν να ζουν σε μουσείο, αλλά θέλουν να έχουν μια αηφόρο ανάπτυξη στην περιοχή τους. και σε ένα άλλο σημείο δεν έρχομαι στο ίδιο αποτέλεσμα όταν ακούω τη λέξη μορατόριο για την εκμετάλλευση των πρώτων υλών. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος ούτε των το πληθυσμών ούτε των αυτοχθόνων ούτε των άλλων των διαφορεμένων όσον αφορά την ε, ακτική γεωργία και την εκτροφή ταράνδων. Ναι, δεν το αναφέρα εγώ έτσι ρητά Ίσως αυτό θεώρησα ότι εντάσσεται στο θέμα της αηφόρου ανάπτυξης των αυτοκτόνων πληθυσμών. Όσον αφορά την βόρεια, την σκανδαλική αυτή διάσταση, η κυρία και το ανέφερε μεταξύ άλλων, ε, πιστεύω ότι η δική μας πολιτική για την Αρκτική δεν θα πρέπει να είναι ε, μια υποομάδα της πολιτικής ε, για την Σκανδιναβία γενικά και την βόρεια περιοχή. Δηλαδή αυτή είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία με ένα παράθυράκι στην Ακτική. Ένας υπουργό της Ρωσίας είχε πει εμείς έχουμε ένα παράθυρο ακτικό, αλλά όχι αρκτική πόρτα. Αυτή η πολιτική της βόρειας διάθεσης είναι δηλαδή μια ε, πολιτική η οποία εστιάζεται κυρίως στη Ρωσία αλλά δεν σχετίζεται και δεν μπορεί να ορίσει την δική μας πολιτική για την Αρκτική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται μόνιμα οι αυτόχθονοι πληθυσμοί, αλλά αυτό για λόγους ε, επικουρικότητας είναι ένα θέμα ε, για την Σουηδία και τη Φιλανδία δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αναλάβει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάνφος Λέζε είπε ότι οι διάφορες πτυχές δεν είναι καλά συνδεμένες μεταξύ τους. Εγώ νόμιζα ότι είχα αναφερθεί ρητά στο ότι αυτές τις διάφορες πτυχές θα πρέπει να τις καταστήσουμε συμβατές. Δηλαδή, αλληλεία... Ε, θαλάσσιες μεταφορές, προστασία των πρώτων υλών, προστασία των, ε, του περιβάλλοντος. Δεν είναι θέματα που αλληλοεξαιρούνται, αλλά θα πρέπει να συνενώσουμε την πολιτική. Έχοντας πάντα κατά ότι δεν έχουμε εκεί κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορούμε να παραποσφέρουμε μια συνεργασία γιατί αν δω ότι τι γίνεται με την Νορβηγία, πώς συνεργαζόμαστε και αναφερόμαστε στα διάφορα ε, συμφέροντά μας για την αλλήλεια, για την ε, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Και τον ίδιο τρόπο που δρά η Ρωσία με την Νορβηγία, πώς χρησιμοποιούνται αυτές τις δυνατότητες, τότε και εμείς σαν ε, εταίρος συνεργασίας μπορούμε νομίζω να συνεργαστούμε. Υπάρχουν δυνατότητε αυτές οι διάφορε πτυχέ να καταστούν συμβατές μεταξύ του. Και έχω εδώ κατά νου το ότι οι κλιματολογικές αλλαγές δεν πρέπει να καταπολεμηθούν μόνο στην Αρκτική, αλλά σφαιρικά και παγκόσμια. Δηλαδή με μονομερή πολιτική στην Αρκτική δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό είμαι και κατά του μορατόριου της εξόριξη των φυσικών πόρων όσον αφορά την ε, σύμβαση με την Αρκτική. Το πρόβλημα είναι ότι στην, ε, στο βορρά εκεί δεν υπάρχουν ελεύθερες γεές, είναι όλα ε, κυριαρχικά κατατεθμημένα. Και δεν μπορούμε να έχουμε κάτι παρόμοιο με την συνθήκη της Ανταρκτικής. Δεν μπορούμε παρά να προσφέρουμε συνεργασία σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς και όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας. Και αυτό αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν θα πρέπει νομίζω να προκαλέσουμε συγκρούσεις γιατί είδαμε καλά αποτελέσματα με την Νορβηγική Ρωσική σύμφαση για τα σύνορα που υπήρχε δυνατότητα σύγκρουσης και δεν έγινε τίποτα. Παραδείγματο χάρη η Νορβηγία αποστέλει παραδείγματο χάρη τις ε, μπαταρίες Στρότσιουμ στους ε, στην ακτή της Ρωσίας. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα που θα μπορούσε να ε, εξεταστεί σαν ένα παράδειγμα σαν ένα παράδειγμα αποφυγής συγκρούσεων. Εάν οι χώρες στην Ακτική έχουν κάποιες βάσεις στρατογικές στη δική τους επικράτεια, μπορούμε εμείς να πούμε δεν επιτρέπεται μπορούμε να προσπαθήσουμε να πούμε ας πούμε διεθνώς να προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν μεγαλύτερες εντάσεις. Ας εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς αυτούς. Και τότε δεν θα υπάρχουν νομίζω συγκρούσεις και εντάσεις. Για την Κίνα είπε ο συνάδελφος ε, ε, Σούλτς ότι θα ήθελε να συμμετάσχει βέβαια να συμμετάσχουν και εκείνοι στην, ε, στο διάλογο και θα μπορέσουμε έτσι νομίζω να υποβάλουμε επικοδομητικές προτάσεις για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε θετικές επιπτώσεις και επικοδομητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της περιοχής. Με χαρά περιμένω τις τροπολογίες σας και τις συζητήσεις που θα έχω και με τους σκιώδεις ηγητές. Θα μπορέσουμε να πούζω να πετύχουμε ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Γκάλερ. Δεν έχουμε άλλες τοποθετήσεις. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 15-11 στις 3 το μεσημέρι. Και η συζήτηση θα γίνει 18 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο. Έκθεση, σχέδιο έκθεσης του Τράιεν Ουγγουρεάνου. Πρόκειται για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα. Το προηγούμενο μήνα είχαμε μια κρόαση σχετικά, όπου εμπειρογνώμονες και συνάδελφοι συνεισέφεραν και τόνισαν ε, την στρατηγική στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας. Ο εισηγητής ήδη έχει προετοιμάσει ένα κείμενο και δίνω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφο Γκουρεάνου. Uh, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στην δημόσια κρέωση, Εκρόαση ε, ε, με συγχωρείτε, εξαιρετικά εμπνευστική και επικοδομητική να εξηγήσω τον περίγυρο και το γιατί αναφερόμαστε στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εύξηνο πόντο. Θα μπορούσα να συνδέσω μάλιστα την έκθεση αυτή με την προηγούμενη, αν και σε πιο ζεστές περιοχές, ακόμα και από στρατηγική πλευρά. Και ακριβώς ένας λόγος η διεκπώνηση αυτής της έκθεσης είναι η ανάγκη ανάπτυξης της πολιτικής για την αντιμετώπιση της κατάστασης ανά τον εύξηνο πόντο. Η έκθεση αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζουμε την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Στο δεύτερο τμήμα διατυπώνουμε προτάσεις για την εδραίωση της δράσης, την αναβάθμιση μάλιστα της δράσης και της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή για να πάρει και τις διαστάσεις μιας πραγματικής στρατηγικής. Η συλλογιστική η οποία μας οδήγησε στην κατεύθυνση αυτή βασίζεται σε διάφορα επιχειρήματα. Καταρχήν, ο εύξηνος πόντος η Μαύρη Θάλασσα, αν θέλετε, έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιδιαίτερα μετά την προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρίας το 2007. Η Μαύρη Θάλασσα εν μέρη είναι από το 2007 εν μέρη επαναλαμβάνω μια εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι τι αλλαγέ που έγιναν το 2007 και το 2008 τις έχετε κατανοήσει. Ήταν η εποχή που και η σχετική πολιτική έκανε τα πρώτα της βήματα στην περιοχή. Τώρα, κατά τα άλλα, πρέπει να αξιολογήσουμε την εφαρμογή αυτής της συνέργειας για τον εύξηνο πόντο να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και τούτο, διότι μεταξύ άλλων δεν υπάρχουν και τα μέτρα και τα μέσα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράση μας. Στον τομέα της εφαρμογή, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λοιπόν εργαλεία παρακολούθησης, αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικείμενο επικρίσεων. Ακριβώς επειδή, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε τρόπο να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της συνέργειας στην περιοχή. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσαμε σχετικά εύκολα να συμπεράνουμε έστω και απουσία μετρήσεων, ότι η εικόνα είναι μεικτή. Φυσικά έγιναν και καλά πράγματα, είχαμε επιτυχίες, κυρίως σε τεχνικά θέματα, στο τεχνικό επίπεδο. Όμως εν γέννη, η εφαρμογή της πολιτικής αυτής έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα, για παράδειγμα, της διακυβέρνησης, της ασφάλειας, τομέα στον οποίο αντιμετωπίζουμε συνεχώς προκλήσεις. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη κατάστρωσης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μαύρη Θάλασσα. θα πρέπει να εδράζεται βεβαίως στην συνεργεία, όμως χρειάζεται ένα καλύτερα δομημένο πλαίσιο πολιτικής. Η πρόταση λοιπόν για την στρατηγική συνδυάζεται άριστα με την στρατηγική ή μάλλον τις στρατηγικές για άλλες μεγάλες περιοχές όπως Βαλτική και ο Δούναβης. Η στρατηγική αυτή λοιπόν στο μέλλον πρέπει πρώτον να εδράζεται σε μια ενιαία οργανωμένη προσέγγιση, πρέπει να περιέχει ένα σχέδιο δράσης καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης, αναφοράς, επισκόπησης, να διαθέτει φυσικά προσωπικό μια γραμμή στον προϋπολογισμό. Και όλα αυτά σε καθεστώς διαφάνειας και τακτικών επαφών με τη μορφή τακτικών υπουργικών συνόδων. Έτσι, θα δώσουμε τέλος στους αποκλεισμούς και θα επιτρέψουμε στους λαούς της περιοχής να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, χωρίς να ξεχνούμε βεβαίω τη σημασία εταίρων όπως η Τουρκία και η Ρωσία. Για να επανέλθω στο βασικό μου μήνυμα, θεωρώ ότι ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή είναι διτός. Ασφάλεια και ενέργεια. Ασφάλεια και ενέργεια. Στο κείμενο, για αυτό το λόγο, Μιλάμε για προτεραιότητες όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, το περιβάλλον, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτά είναι οι προτεραιότητες μας. Και για να μην μακρηγορώ. Φυσικά πρόκειται για ένα ε, σχέδιο. Το σχέδιο όμως της έκθεσης περιλαμβάνει σίγουρα τα βασικά σημεία. Θα προσπαθήσω να εμπλουτίσω αργότερα το κείμενο χάρη και στις ε, τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και δι τους σκιώδεις ε, εισηγητές καθώς και τους ε, αρμοδίους για τις γνωμοδοτήσεις και βέβαια τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι όλος αυτιά για σχόλια και απόψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σούλτ, σκιώδη εισηγητή. Bericht zur eu schwarzmeer strategie geht von den Schwerpunkten und den Zielsetzungen. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μαύρη Θάλασσα έχει ορισμένα κενά που θα πληρωθούν, ελπίζω, μέσα από τις τροπολογίες. Και έχω τρεις εδώ. Δημοκρατία και κοινωνία των πολιτών. Αν θέλουμε να τις προθίσουμε πραγματικά, πρέπει να ενισχύσουμε τα διασυνοριακά δίκτυα. Πριν από 20 χρόνια έπεσε το τείχος και δεν θα σταματήσουμε εμείς να επιμένουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία διασυνοριακών δικτύων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σαφώς να τα χρηματοδοτεί όλα αυτά τα σχέδια. Χρειάζονται επίσης συστήματα έγκαιρου συναγερμού Λόγω της ε, συνοχής παρουσίας ε, της ρωτοριστικού ε, στόλου της Μαύρης Τρίτων μια τροπολογία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας ε, δημοσιακά και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Και αυτό θα πρέπει να προσθέσει σε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκόβατσεκ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βουλιάνοφ για το σχέδιο έκθεσή σα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία τη έκθεση αυτή και θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μια στρατηγική για την Μαύρη Θάλασσα, καλύτερο συντονισμό. Δεν αναγνωρίζεται ακόμα επαρκώ η στρατηγική σημασία για το εμπόριο, την ενέργεια, την ασφάλεια και τι μεταφορέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια νέα ισχύ στην περιοχή αυτή και θα πρέπει να αυξήσει την παρουσίασή τη και πολιτικά και οικονομικά πολιτικά με την υποστήριξη των χωρών στην περιοχή εκεί για να εξελιχθούν πιο ε, δημοκρατικά και να εφαρμόζουν καλύτερα το κράτος δικαίου. Θα πρέπει επίσης να ε, έχουμε υπόψη τις παγωμένες και τόσο όχι τόσο παγωμένες συγκρούσεις της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι κύριος συμμετέχοντας στη δημιουργία καλύτερη συνεργασίας περιφερειακά και καλύτερου περιφερειακού εμπορίου. Θα πρέπει εκεί να δούμε την διαμεθοριακή συνεργασία. Καλό αυτό, αλλά δεν βασίζεται στις προσδοκίες μας απόλυτα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα πιο σκληρό ρόλο στην ασφάλεια της ε, περιοχής της ε, Μαύρης Θάλασσας. Ιδίως θα πρέπει να περιοριστεί η διεύρυνση των εξοπλισμών και να περιοριστεί το λαθρεμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες διαχωριστικές ε, γραμμές γιατί στην Μαύρη Θάλασσα έχουμε πολλές τέτοιες γραμμές και τελευταία είδαμε καινούριε ιδίω στον Κάφκασο. Θα πρέπει να εργαστούμε για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον με τη δημιουργία ειρήνης και εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να αποφύγουμε η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οδηγήσουν σε αύξηση των συγκρούσεων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ειρηνικέ επιλύσεις. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σε λύση στις προκλήσεις της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισχύς με παγκόσμιες προδοξίες θα πρέπει να φροντίσει να διευκολύσει εκεί την διαμεθορική συνεργασία και το εμπόριο. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της περιοχής που ανέφερε ο κ. Κιγκουρεάνος στην έκθεσή του και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το διοικητικό της δυναμικό και η υπηρεσία, η μελλοντική της εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει επαρκή δυναμικό για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ηγέτη στην περιοχή. Όπως και οι συναδελφοί και εγώ ζητώ να υπάρχει ένα άλλο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και καλώ την ε, να συνεργαστεί σε μια πλήρη στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα που θα βασίζεται στις περασμένες εμπειρίες της ε, περιοχής. Ένα συγκεκριμένο μέτρο που θα ήθελα να εφαρμοστεί στην ε, Μαύρη Θάλασσα είναι ο συντονισμός των ε, δράσεων αναζήτησης και διάσωσης. Είχαμε ένα πολύ άσχημο παράδειγμα με ένα ε, πλοίο που να ναυάγησε όχι πολύ μακριά από την, ακτική, από την ακτή. Συγγνώμη. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ε, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ πλούσια. Αυτό δυστυχώς δεν είναι καλά γνωστό και γι' αυτό Πιστεύω ότι στην περιοχή της ε, Μαύρης Θάλασσας θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα που θα προωθούν την πολιτιστική ανταλλαγή και θα προωθούν και τον τουρισμό. Και ελπίζω αυτό το θέμα να μην ενδιαφέρει μόνο τους Ρωμάνους και Βουλγάρους μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και τα άλλα μέλη από άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε τοποθετήσεις και την απάντηση του εισηγητή στη συνέχεια. Παρακαλώ λοιπόν να είστε πιο σύντομοι ως η συνάδελφος Νικολάη, τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση αυτή και να αναφερθώ στην αποτελεσματικότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γιατί και το 2007 Ξεκινήσαμε με ένα θέμα συνέργεια τη Μαύρη Θάλασσα και μέχρι στιγμή δεν έγινε τίποτα. Θυμάμαι και την ανατολική εταιρική σχέση που δεν είναι σε πολύ καλή θέση εντό Και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι ένα ε, σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, ιδίως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής μας γυτνίασης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα που αναφέρουν στην σημασία της πολιτικής αυτής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Γιατί θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ καλά για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιφερειάς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την διανυστρία τόσες διαμάζες που υπάρχουν Αζερβαϊτζάν και άλλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπλακεί και, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ε, να εμπλακούμε ακόμα περισσότερο στην δράση στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν διάφορα σημεία που θα πρέπει νομίζω να αναφερθούν. Ε. Καταρχήν το θέμα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την μετανάστευση, μιλάμε για την ασφάλεια των συνόρων, και πρέπει να δράσουμε γιατί εκεί έχουμε ε, μια πύλη για τους μετανάστες που έχουν από την Ασία και θα πρέπει γι' αυτό η ασφάλεια των συνόρων να αυξηθεί. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στο εμπόριο ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση και το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών βέβαια σημαντικό, αλλά κυρίως και το λαθρεμπόριο των ανθρώπων. Πιστεύω ότι η στρατηγική θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό θέμα και στις ε, νέες σχέσεις με τη Ρωσία. Γιατί αναφερόμαστε στο θέμα των σχέσεων Ευρώπης-Ασίας και η ε, Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικό τμήμα των σχέσεων αυτών. Ευχαριστώ. Κολίγα Κύριλοφ you have the floor. Ο συνάδελφος Κυριλόφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω στα προηγούμενα σχόλια ότι βεβαίω προσπαθούμε τώρα να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην περιοχή του Ευξηνού Κάτι το οποίο όμως ήταν δύσκολο ως τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε εν πάση περιπτώσει κάτι επιτέλους και ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε με αποτελέσματα γιατί αλλιώς όλα αυτά θα παραμείνουν ευθεβείς πόθη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί, όπως είπαν και άλλοι, με την Βουλγαρία και την Ρουμανία, μέλη της υπερχής Σέγγεν, κάποιοι θα εστιάσουν τη δική τους προσοχή στην περιοχή από την άποψη του εμπορίου ανθρώπων όπως έγινε και με την Μεσόγειο. Λοιπόν, αν δεν δώσουμε επαρκή προσοχή στο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα προβλήματα. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων και θα χρειαστεί να εμπλέξουμε και την πολιτική για τον Δούναβη εκτό από την Μαύρη Θάλασσα. Γιατί στην περιοχή, εκτό από τον εμπόριο ανθρώπων, θα αντιμετωπίσουμε και θέματα που άπτονται τη τρομοκρατία. Γιατί τα δύο αυτά, όπω ξέρετε, είναι αλληλοσυνδεόμενα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι πτυχέ τη στρατηγική. Στον τομέα όμω ειδικότερα τη ασφάλεια, τη στρατηγική, του προπολογισμού, χρειαζόμαστε να είμαστε πρακτικοί για να έχουμε αποτελέσματα να πετύχουμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να δείξουμε ειδικό ενδιαφέρον, αλλιώς θα παραμείνουμε στο πλαίσιο της παλιάς συνεργεια Χατζη εγω Εγώ έχω μια-δυο σκέψεις και ίσως ταυτόχρονα να είναι ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Χωρίς αφιβολία είναι μια κρίσιμη περιοχή για τον κόσμο, πολύ περισσότερο κρίσιμη περιοχή για τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες. Εγώ δεν κατάλαβα, υπήρξε μια κοινή σύσκεψη ή μερικές κοινέ συσκέψεις των κυβερνήσεων των χωρών που έχουν να κάνουν με τη Μαύρη Θάλασσα για να δούμε τι εισηγήσει έχουν ήδη για την περιοχή τους. Πολύ περισσότερο ο εισηγητής ή και από μόνα τους τα κοινοβούλια των χωρών που έχουν να κάνουν με τη Μαύρη Θάλασσα είχαν κάποιου τύπου κοινέ συζητήσει για το κοινό τους μέλλον γύρω από την ε, δική τους ε, θάλασσα. Ε, θέλω να πω να μην φαίνεται ή και να μην είναι δηλαδή μια παρέμβαση ή η παρεμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια που να μην ουσιαστικοποιεί την συμμετοχή των εκπροσώπων των, των λαών στην περιοχή και αναφερόμενος σε λαούς έρχομαι πάνω στο, στο κυρίως θέμα που θα ήθελα να, καταθέσω. Ε, ασφάλεια και ενέργεια, είπε ο εισηγητής, είναι ε, τα κύρια ζητούμενα και χωρίς αμφιβολία ε, είναι πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Από τους επόμενους ομιλητές μπήκε και το θέμα της μετανάστευσης. Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχουν ε, πολίτες, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ε, δύσκολα ή πολύ πιο δύσκολα τη ζωή τους. Το ερώτημα είναι μέσα από την εισήγηση ή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπαίνουν σε τροχιά στρατηγικές σκέψεις που να βγάζουν τον κόσμο της περιοχής αυτής από την φτώχεια ε, έτσι ώστε η αηφόρος όπως την λέμε η ανάπτυξη να είναι κυρίως δουλειά δική τους και να μην ε, προάγει ε, και την μετανάστευση η οποία φυσιολογικό είναι να υπάρχει όταν οι άνθρωποι στους τόπους τους ε, έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και θεωρούν ότι η μετακίνησή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους δώσει καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ. Grazie. Ε, la parola al collega Preda, prego. Ο συνάδελφος Πρέντα. Πρόεδρε, συγχαρητήρια καταρχήν στον συνάδελφο για το κείμενο. Δεύτερον, θα ήθελα να συνηγορήσω με την εξαιρετικά πιστική έκκληση που διατυπώνεται εδώ σχετικά με την στρατηγική σημασία του ευξήνου πόντου. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα τονιστούν περαιτέρω και κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης που θα ακολουθήσει το τελικό κείμενο, μετά βεβαίως και από την κατάθεση των τροπολογιών. Από πολιτικής απόψεως, Έχει σημασία να τονίσουμε την στρατηγική σημασία του ευξήνου πόντου. Και τέλος, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο εισηγητής έχει απολύτως δίκιο όσον αφορά τα σχολιά του στο προήμιο. Εκεί που τονίζει δηλαδή ακριβώς την αποσπασματική προσέγγιση της πολιτικής μας για την περιοχή αυτή ως τώρα και η τρέληψη των σχετικών πόρων. Θα έπρεπε να είχαμε χρηματοδοτήσει ένα, για παράδειγμα, πιλωτικό πρόγραμμα για την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Ξέρω ότι κάποια χρήματα είχαν πρικοδοτήσει μια προσπάθεια, αλλά τελικώς χρησιμοποιήθηκαν για άλλη περιοχή. Η αποσπασματική λοιπόν αυτή χρηματοδότηση τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια αυτών που προσπαθούν για τον εύξηνο πόντο. Ας κάνουμε λοιπόν εμείς ως βουλευτές ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ο παρέμβαση, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και συγγνώμη που άργησα. Δυστυχώς με καθυστέρησαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Καθυστέρησα και με μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Ουγγουρεάνου για ένα εξαιρετικό κείμενο. Πιστεύω ότι η ανάλυση του εισχώρησε σε βάθος και δεν υπάρχει λόγος να παραλάβω τα όσα είπαν οι προελίσσαντες. Βεβαίως είναι σημαντικά αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η περιοχή αυτή συνδυάζει την παρουσία πολλών χωρών. Δεν έχουν όλες την ίδια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μερικές από τις χώρες της περιοχής έχουμε επαφές. Κάποιες χώρες επίσης διαδραματίζουν ούτως ή άλλως σημαντικό ρόλο στην περιοχή και περιμένουν και το δικό μας επικοδομητικό ρόλο. Ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, να στήσουμε την άποψή τους, να, τις, να τους επιτρέψουμε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δικής μας στρατηγικής. Στρατηγικής η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Πιστεύω ότι αξίζει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για την κατάστρωση αυτή τη στρατηγική, η οποία με τη σειρά τη θα συμβάλλει στην σταθερότητα στην περιοχή. Πρόκειται για όμορη περιοχή προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λανθάνουσε συγκρούσει στην περιοχή, οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να επεμβαίνουμε έγκαιρα όπου χρειάζεται να συνδράμουμε επίσης στην εξέβρεση λύσεων. Η περιοχή αυτή είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως λέει άλλωστε και η έκθεση, από ενεργειακής απόψεως, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Αυτό το οποίο έχει πλέον μεγάλη σημασία κατά την απόψή μου είναι η στρατηγική να εστιαστεί και στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών και δημοκρατικών κοινωνιών και καθεστώτων στην περιοχή και ιδιαίτερα στις χώρες και τις περιοχές που έχουν βλέψεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. Μην ανησυχείτε για την καθυστέρηση. Ε, ο Δόκτωρ Πέσσε. Επιτρέψτε μου εισαγωγικώς να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή το κείμενο είναι ουσιαστικό, εμπεριέχει πολλές ιδέες, αναφέρεται και στο μέλλον αλλά και στις παρούσες προσπαθίες μας με τρόπο ισορροπημένο. Πιστεύω ότι βάσει του κειμένου θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε σύντομα περισσότερα. Να υπενθυμίσω απλώς ότι η συνεργία για την ε, Μαύρη Θάλασσα είναι ένα απλώς από τα στοιχεία της πολιτικής μας για την περιοχή. Γιατί έχουμε πολιτικές ε, με τα, κείμενα, κράτη της περιοχής, έχουμε σχέσεις, βαθιές σχέσεις και όλα αυτά είναι τίματα της στρατηγικής. Η συνέργεια λοιπόν συγκυράζει τα κοινά στοιχεία, τα στοιχεία της εργασίας αυτής της πολιτικής. Δεν θα σχολιάσω όλες τις κρατάλα αλλά πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Θα μελετήσουμε όλες τις προτάσεις πολύ προσεκτικά. Φυσικά θα προκύψουν κάποιες προτεραιότητες όπως η ασφάλεια, όπως η μετανάστευση. Πρόκειται για θέματα τα οποία θα αποτελέσουν μέρος φυσικά της στρατηγικής και των περαιτέρω ενεργειών μας. Πολύ σύντομα, επίσης, να πω ότι δεν μπορούμε να υποτιμούμε τις δυσκολίες υλοποίησης του όλου εγχειρήματο. Η περιοχή είναι δύσκολη, να μην αναφερθώ στις συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά να υπενθυμίσω τουλάχιστον ότι ως τώρα προσέγγισή μας από τεχνικής απόψεως είναι μια βήμα προς βήμα τακτική. Και αυτό αντικατοπτρίζει ακριβώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ακόμα και σε τεχνικό επίπεδο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πέρα λοιπόν από τις ε, δυσκολίες εφαρμογής, δεν υπάρχει καμία εμφολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχους στη Μαύρη Θάλασσα. Θα έλεγα ότι ο ισχύτης θα δικούσε αυτόν εάν τις δυσκολίες αυτές, τις πρακτικές δυσκολίες, θα, θα τους επέτρεπε να περιορίσουν το πολιτικό μας όραμα και το οποίο είναι ένα σαφές πολιτικό όραμα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ε, για να κάνουμε και τη συζήτηση πιο ενδιαφέρουσα, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις η την υλοποίηση του εγχειρήματο και όχι μόνο πολιτικέ. Η εμπλοκή, η άμεση εμπλοκή καταρχήν των χωρών στην περιοχή, αλλά και πολύ πιο κοντά μα αν θέλετε. Υπάρχουν διοικητικέ, οικονομικέ, χρηματοδοτικές προποθέσει, Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να διαδραματίσουμε ρόλο στην περιοχή, πρέπει να αναλάβουμε και το κόστο. Τόσο απλά. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιονομικές υποχρεώσεις, αλλά και υποχρέωση εμπλοκής πόρων, ανθρωπίνων και άλλων. Ε, γι' αυτό θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες. Αν υποσχεθούμε κάτι, να πούμε και πώς θα το υλοποιήσουμε. Όπως άλλωστε ένας βουλευτής το υπενθύμησε, η δημιουργία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι μια χρυσή ακριβώς ευκαιρία για να προσδιορίσουμε την εμπλοκή μας στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δ. Μπεσέ, για την σαφήνεια με την οποία μιλήσετε Ο εισηγητή για τα συμπεράσματα, παρακαλώ. Ο κ. Τραγιάν Ουγγουριανού Πρόεδρε, ήδη είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Κατέθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλια και απόψει. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μάλλον Ήδη συμφωνούμε ως προς την στρατηγική σημασία της περιοχής. Συμφωνώ με όλους. Δεν πρόκειται για ελληνο-ρουμανο-βουλγαρική υπόθεση. Ακόμη και αν αυτό ενδεχομένως ίσχυε στο παρελθόν, σίγουρα η περιοχή ενδιαφέρει την Ευρώπη συνολικά. Δεν πρόκειται λοιπόν για περιφερειακό ζήτημα με τα συν και τα πλήν του. Ο κ. Σούλτς ορθότατα υπογράμμισε τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Μίλησε για το εμπόριο ναρκωτικών. Ο κ. Σκοβάτσεφ επίσης ε, ορθώς αναφέρθηκε στα όπλα, στα ναρκωτικά και τα σχετικά προβλήματα θα ενσωματώσω την παρατηρήσή του. Το ανέφεραν άλλωστε και άλλοι ομιλητές. Είναι επίση σωστό ότι δεν υπάρχει διμερή λύση, αν θέλετε, για τα σχετικά προβλήματα. Κύριε Κόβατσεφ, έχετε δίκιο ω προ τον κατεπήγοντα χαρακτήρα επίλυση των θεμάτων έρευνα και διάσωση στην Μαύρη Θάλασσα. που δυστυχώς τους δύο τελευταίους μήνες ε, έγιναν εξαιρετικά επίκαιρα. Δεν κύριε Ρεκολάη, συμφωνώ. Στο πλαίσιο της συνέργειας για τον εύξηνο πόντο δεν έγιναν πολλά. Ο κ. Μπεσέ πάντως ε, είχε δίκιο. Είπε ότι η συνέργεια δεν είναι μόνη μας πολιτική. Απ' την άλλη πλευρά, ας μην υποτιμήσουμε τις δυνατότητες Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση ευκαιρίες αλλά και δυσκολίες. Επίσης, ε, σύμφωνα με τον κύριο Κύριλοφ, έχει δίκιο όταν λέει ότι η περιοχή θα γίνει ακόμη πιο σημαντική για την Ευρώπη όταν Ρουμανία και Βουλγαρία γίνουν μέρος της ζώνης Σέγγεν. Δεν θέλουμε η περιοχή να μεταβληθεί σε μια νέα Μεσόγειο. Από την άποψη της μετανάστευση. Και προς τον κύριο Χατζηγεωργίου φυσικά χρειαζόμαστε μια ανοιχτή κοινή συζήτηση. Έγινε αυτό στο Κίεβο σε υπουργικό επίπεδο το 2008. η συζήτηση αυτή, ο διάλογος αυτός, ο μηχανισμό αυτός σίγουρα πρέπει να επαναδρομολογηθεί, να επανακινητοποιηθεί. Και κύριε Πρέντα, μίλησατε και πάλι για την στρατηγική σημασία τη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, όπως φαντάζεστε, σύμφωνα απολύτως. Και ο κ. Σμάκεν μίλησε για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σαφώς πρέπει να το δούμε και θα το συμπεριλάβω στο σχέδιο και εν τέλει στο τελικό κείμενο. Ως προς τα όσα είπε ο Δ. Μπεσέ από την Κομισιόν, Δόκτωρ Μπέσε, η ανάλυση ε, ήταν εξαιρετική όσον αφορά τα ειδικά πολιτικά χαρακτηριστικά της περιοχή, τα ειδικά στρατηγικά χαρακτηριστικά τη περιοχή, ε, κάτι το οποίο δεν κάνει τη ζωή μα, ε, θα λέγα, εύκολη στον εύξηνο πόντο. Όπως είπε ο δόκτωρ Μπεσέ, δεν έχει τελειώσει η δύσκολη περίοδος Παιδίζουμε ακόμη σε λασπόδες έδαφο. και σίγουρα χρειαζόμαστε χρήματα. Αν θέλουμε να διδραματίσουμε ρόλο στην περιοχή, πρέπει να πληρώσουμε και να δείξουμε μια στάση συνεπή, μεταξύ άλλων και οικονομικός συνεπή. Αυτά προς το παρόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρος. Να μην ξεχάσω να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των είναι 12 η ώρα 16 Νοεμβρίου 16 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε εδώ γιατί ακολουθεί το διευρυμένο Προεδρείο το οποίο θα συνεδριάσει